Τίμιο Παλατσκι αναπτύσσει μια εφαρμογή για γονεί και παιδιά μπορούν να αξιολογήσουν έτσι καλύτερα του κινδύνους. Αυτό χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ναι, με μικρόφωνο. Ε, Τσόχονταρ από του σοσιαλιστέ και δημοκρατε. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα παιδιά ε, συνεχίζουν να είναι ευάλωτα και έχουμε πολλές ανησυχίες, ειδικά όσον αφορά το περιεχόμενο που κυκλοφορεί online, παιδική πορνογραφία, παιδοφιλία, bullying, ε, εκβιασμοί. Επίσης υπάρχουν κίνδυνοι όσον αφορά τη δυνατότητα της χρήσης του ίντερνετ. Εγώ στα παιδιά στην πόλη μου που είναι ε, προσχολημένα στο ίντερνετ, που έχουν αναπτύξει κάποιες παθήσεις επειδή ε, βρίσκονται μπροστά στις οθόνες υπερβαλικά πολύ χρόνο ε, πρέπει να υπάρξει μέρημνα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση και το ίντερνετ να είναι ασφαλές, ασφαλής χώρος. Ποια είναι τα τρία μέτρα που προτίθεστε να πάρετε καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφος Περέιρα από την ΚΟΕ. Το ίντερνετ για τα παιδιά υπάρχουν κίνδυνοι παραβίαση της ε, προσωπική ζωής, κίνδυνοι για την υγεία και εμφάνιση φαινομένων εξάρτησης ε, και απώλειας ε, της ταυτότητας. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τα, την σεξουαλική παρενόχληση, τα τυχερά παιχνίδια αλλά και την ακατάλληλη διαφήμιση, τη βία, το σεξ και άλλες καταστάσεις που φοβίζουν τα παιδιά. Είναι απαραίτητο να εγγυηθούμε τα παιδιά να εκτίθεται όσο γίνεται λιγότερο σε αυτός τους κινδύνους. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας όσον αφορά μέτρα που μπορεί να ληφθούν χωρίς να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Επίσης, θεωρούμε πως αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη σημασία της δημόσιας ε, ε, υπηρεσίας, την εγγύηση της ασφαλούς υπηρεσίας και της καθολικής υπηρεσίας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Επίτροπος Ντάλη τώρα. Σας ευχαριστώ όλους για τις ε, συμβολές σας. Σημείωσα όλα σας τα σχόλια σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ανέφερα, τα ανέφερα ήδη ε, στην εισήγησή μου. Πριν ε, δηλαδή να αρχίσετε εσείς να σχολιάζετε η Κομισιόν με χαρά βλέπει πως το θέμα αυτό παραμένει υψηλή προτεραιότητα και είμαστε πεπισμένοι ότι νέα μέτρα στο τομέα αυτό θα βρουν την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο μπορεί να βασιστεί στην πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, μάλλον ότι θα προωθήσουμε την ασφάλεια, ε, την επιγραμμική ασφάλεια των παιδιών. Εμείς θα ε, προσπαθήσουμε πάντοτε υπέρ της προστασίας των παιδιών με υψηλές προδιαγραφές προστασίας και ε, θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε την, τον κλάδο ολόκληρο γιατί τα σημερινά παιδιά θα είναι οι αυριανοί ε, υπεύθυνοι πολίτες και γι' αυτό και θα πρέπει να τους προστατέψουμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτές για τη συμβολή σας σε αυτή τη συζήτηση. Και όπως είπα ήδη έχω σημειώσει όλες σας τις ε, παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή και περνάμε στο τελευταίο θέμα για τη σημερινή μας ημερήσια διάταξη. Κορονοϊός. Διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση. Και πάλι θα σας δώσω το λόγο, κυρία Ντάλι, εξονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Possible only after the group's opinions, okay? Thank you. So, thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. ναι προφανές ότι είναι τεράστιες προκλήσεις για από την αύξηση της αντιμικροβιακής ε, αντίστασης ε, και ε, μαζί με την κλιματική αλλαγή οι απειλές αυξάνονται. Ο, αυξάνονται. ο κορονοϊός είναι απόδειξη αυτού και δείχνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκτός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας σημαντικός σύμμαχος και εταίρος σε αυτή την προσπάθεια και χαίρομαι που θα συζητήσω μαζί σας την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινητοποιήσει τις υπηρεσίες της, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων για παράδειγμα, προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών να αντιμετωπιστεί ε, η ε, κατάσταση. Συνεργαζόμαστε και συντονίζουμε τη δράση μας με τα κράτη-μέλη, ε, χρηματοδοτούμε εμβόλια και στηρίζουμε τα κράτη-μέλη με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Θα σας δώσω παραδείγματα από τις προσπάθειές μας και ιδέες για μια βελτιωμένη ανταπόκριση. Αλλά καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω και να συγχαρώ όλο το ιατρικό προσωπικό πρώτη γραμμή ε, που εργάζεται σε πολύ δυσχερή συνθήκες. Την περασμένη εβδομάδα εκφράσαμε τα συλληπιτήριά μας ιδιαίτερα για τον θάνατο του δόκτρος Λου Λου Λάγκ που ήταν μεταξύ των πρώτων που μας προειδοποίησε για την επικίνδυνοτητα του ιού. Ε, μερικά λόγια για την σημασία του συντονισμού μεταξύ διαφόρων τομέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις 26, 28 Ιανουαρίου η πρόεδρος Φάντερ Λάγεν ε, ε, συγκάλεσε το μηχανισμό το συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ε, Επίτροπος ε, διορίστηκε ως επικεφαλής του μηχανισμού και προείδρευσε αυτού με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών της ε, Κομισιόν, υγείας, πολιτικής προστασίας, έρευνας, μεταφορών, αλλά και αναπτυξιακής συνεργασίας και επικοινωνίας, επικοινωνιών. Συγγνώμη. Ε, επανέλαβε ότι αυτή η πρόκληση απαιτεί μια συλλογική προσπάθεια και τη χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτουμε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Κομισιόν αξιολογούν συνεχώς και τακτικά την κατάσταση και αποφασίζουν για τις απαραίτητες δράσεις ε, προκειμένου να δοθεί κατάλληλη και γρήγορη απάντηση συνεργασία και ο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση επίση συνεχίζεται προκειμένου να επαναπατριστούν πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπιστούν άλλε προξενικέ ανάγκε. Χάρη στο μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολιτική προστασία και, και την προσπάθεια χαρών όπω η Γαλλία και η Γερμανία, εκατοντάδε Ευρωπαίοι πολίτε επαναπατρίστηκαν από την Κίνα. Η Επίτροπος κυρία Κυριακίδου είναι σε τακτική επαφή με, τα, με τους υπουργούς των κρατών μελών ε, που έχουν ε, πληγεί. Η Κομισιόν συντονίζει ε, τα κράτη-μέλη μέσω τριών προμηχανισμών. Τον, το σύστημα γρήγορης έγκαιρης προειδοποίησης, την Επιτροπή Υγείας και το δίκτυο επικοινωνίας. Η, η αποτελεσματική συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη. Οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν σωστά, ανταλλάσσουμε πληροφορίες ε, και διαμορφώνουμε στρατηγικές. Ε, ταυτόχρονα η Κομισιόν χρηματοδότησε με 10 εκατομμύρια ευρώ ε, την έρευνα για τον κορονοϊό. Το πρόγραμμα PREPARE ε, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει κλινικές δοκιμές σε 3.000 νοσοκομεία και 900 εργαστήρια σε, όλη την, σε όλο τον κόσμο, 42 χώρες, ε, έχει ενεργοποιηθεί. Επίσης, ε, συστήσαμε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στα σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα κράτη-μέλη χρειάζεται να, να επεξεργαστούμε μια κοινή στάση στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τις διεθνείς ε, συστάσεις προστατεύοντας ταυτόχρονα και την ελευθερία κυκλοφορίας των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε και να συντονίσουμε τη δράση μας με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους διεθνείς ε, οργανισμούς. Ε, θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ε, το σχέδιο προετοιμασίας ε, για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού μέσω και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ε, η δράση μας είναι ιδιαίτερα σημαντική σε χώρες που έχουν ευαίσθητα συστήματα υγείας. Η Κομισιόν εξετάζει τις ανάγκες των κρατών μελών. Εν παράλληλα, ε, εξετάζει το ποιες είναι οι ικανότητες των κρατών μελών για θέσεις σε καραντίνα. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας στα κράτη-μέλη και διαφορετικές ε, ικανότητες, ε, διαφορετική αριθμή προσωπικού. Χρειάζεται λοιπόν να δειχθεί διασυνοριακή αλληλεγγύη και συνεργασία. Είναι σημαντικό να περιοριστούν τα κρούσματα, να περιοριστούν οι πιθανότητες περαιτέρω διάδοσης του κορονοϊού και, να, και πρέπει γι' αυτό να ε, ε βοηθήσουμε την ίδια την Κίνα. Βοηθάμε την Κίνα και ταυτόχρονα βοηθάμε και εμά του υπόλοιπου όλων τον κόσμο. Η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με την Κίνα σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη παράσχει 12 τόνους προστατευτικού εξοπλισμού στην Κίνα. Αυτό δείχνει πόσο αλληλέγγυοι είμαστε. Είμαστε σε επαφή με ιδιωτικέ εταιρείε και με κράτη-μέλη προκειμένου να εντοπίσουμε πού υπάρχουν αποθέματα τέτοιου εξοπλισμού ε, που ε, δεν τα χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να τα μοιραστούμε με την Κίνα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκή απαθώματα σε εθνικό επίπεδο. Αλλά πρέπει να δούμε και πού η υποστήριξή μας θα είχε τα καλύτερα και τα πιο ε, χρήσιμα αποτελέσματα. Θα δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασία μεταξύ εμπειρογνωμών Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα για τι πτυχέ που έχουν σχέση με την υγεία ε, και τον ιό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις έμεσες συνέπειες του ιού. Για παράδειγμα, η πιθανότητα δημιουργίας φαινομένων ξενοφοβίας ε, διαδικτυακά και στον πραγματικό κόσμο. Η διακρίση εναντίον των Ασιατών ή ατόμων που θεωρούνται ότι είναι Ασιάτες ε, ή οποιασδήποτε άλλες διακρίσεις με βάση την εθνοτική προέλευση είναι αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο και η Κομισιόν δεν θα δεχτεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Η Κομισιόν είναι σε επαφή με την Υπηρεσία Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις ε, αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για να εκτιμήσει την κατάσταση ε, των ε, δραστικών ουσιών που είναι απαραίτητες για την Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία και τελικά την Ευρωπαϊκή Αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει επηρεαστεί η διαθεσιμότητα φαρμάκων στην Ευρώπη, αλλά θα παραμείνουμε σε γρήγορση. Είναι προφανής η ανάγκη όμως να εξετάσουμε την ε, ε, ευρωπαϊκή παραγωγή αντιοικών φαρμάκων. Θα, το αποτέλεσμα θα μας ε, δώσει στοιχεία για την φαρμακευτική στρατηγική την οποία θα ξεκινήσουμε αργότερα φέτος. Ε, εμείς ενεργοποιούμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε και όλο το προσωπικό που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Η επιτυχία μας εξαρτάται από την γρήγορη επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών, την πολιτική βούληση και, την στενή, και το στενό συντονισμό. Όλες αυτές οι προσπάθειες χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη μεταξύ όλων των Ευρωπαίων πολιτών και άλλων πολιτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ευάλωτοι. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω τον λόγο τώρα στην ε, κυρία Ντελάγκη από το ΕΛΚΝΕ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύρια Επίτροπε, αύριο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Υγείας ε, και νομίζω πως είναι πολύ σωστό το ότι συζητάμε αυτό το θέμα απόψε και να είμαστε σαφείς. Δεν χρειάζεται πανικός, δικαίως ο κόσμος ε, στρέφεται στις εθνικές αρχές αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν τις προσπάθειες συντονισμού. Σε προηγούμενες φορές ε, δεν υπήρχε συντονισμός. Εδώ πέρα όμως υπήρξε συντονισμός ε, για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων υπηκών. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο οι υπουργοί αύριο θα τονίσουν ότι η υγεία είναι εθνική αρμοδιότητα και θα έχουν δίκιο όλα ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να μιλήσει για τη συνθήκη της Λισαβόνας, θέλουν λύσεις. Άρα από το ΕΛΚ εμεί περιμένουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα έλεγχος ικανοτήτων όσον αφορά την ετοιμότητα κατώμενων και ανησυχώ όταν η Κομισιόν λέει μπορεί να χρειαστεί να οργανώσουμε την αλληλεγγύη για τον προστατευτικό εξοπλισμό. Όχι. Πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να το τσεκάρουμε. Μια κοινή προσέγγιση επίσης για όσους έρχονται από αυτή την περιοχή και μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, ξεκάθαρη επικοινωνία γιατί βλέπουμε αντικρουόμενες οδηγίες. Για το εμβόλιο τα είπατε, αλλά τέλος επίκαιρα δεδομένα. Πώς είναι δυνατόν να λέμε επισήμως η Αφρική δεν έχει κανένα κρούσμα είτε ε, δεν έχουν κανένα κρούσμα, αλλά είναι λίγο απίθανο δεδομένων των επαφών με την Κίνα, ή δεν ελέγχουν. Αυτό όμως είναι ανησυχητικό, γιατί εμείς ε, είμαστε γειτονική ήπειρος. Πρέπει λοιπόν οι Υπουργοί να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αδύναμοι κρίκοι καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γκούτελαντ από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ και για την ε, σημαντική παρουσίασή σας. 40.000 ε, επιβεβαιωμένα κρούσματα, πάνω από 1.100 θάνατοι. Ε, πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά τον κορονοϊό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα κρούσματα στην Ευρώπη δεν ήταν τόσο πολλά, αλλά η ετοιμότητα είναι σημαντική. Ο Παγκόσμιο οργανισμό Υγεία ε, προσπαθεί να αντιληφθεί ε, το τι γίνεται και η δουλειά του είναι πάρα πολύ σημαντική. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς μεταδίδεται. χαίρομαι επίσης που αναφέρατε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα επί του ιού που νομίζω θα είναι αποφασιστικές η δουλειά που κάνουν οι ομάδες ε, των ειδικών για να βρουν την ε, πηγή της επιδημίας και για να προλάβουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, δεν ξέρουμε αν κάνουμε αρκετά και δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε αρκετά μέχρι να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για τον ιό και το πώς λειτουργεί. Λοιπόν, απευθύνω έκκληση στους Υπουργούς Υγείας να είναι έτοιμοι να δράσουν σε περίπτωση νέων κρουσμάτων και να φροντίσουν να διαδοθούν οι πληροφορίες στο κοινό. Μέτρα για να προλάβουμε την διάδοση του ιού είναι πάρα πολύ σημαντικά και η καραντίνα επίσης ε, των ε, υπόπτων ασθενών ε, είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να γίνεται με τρόπο αναλογικό. Πρέπει να φροντίσουμε επίσης ο κορονοϊός να μην οδηγήσει σε διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τούτων λεχθέντων όμως είναι θετικό το ότι η Κομισιόν ασχολείται με το ζήτημα και είστε εδώ σήμερα για να μας πείτε ότι υπάρχει ετοιμότητα και όλοι μαζί ε, θα διασφαλίσουμε ότι ε, υπάρχει η τεχνογνωσία και θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Τσεχ για το Ρήνιο. Έχετε τον λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε μια μέρα δεν περνάει χωρίς να έχουμε καινούργια νέα για τον κορονοϊό και ο κόσμος κρατάει την ανάσα του και περιμένει να ξεσπάσει μια παγκόσμια πανδημία. Ψευδείς ειδήσει κυκλοφορούν πολύ παραπλανητικές. Στην Ουγγαρία δύο άνθρωποι κρατήθηκαν ε, μετά από ψευδείς ειδήσει στα κοινωνικά μέσα για εκατοντάδες, ε, για μόλυνση μάλλον, με εκατοντάδων ανθρώπων, ανοησίες δηλαδή. Έπειτα 60% λέει της ανθρωπότητας ε, θα μολυνθεί στο μέλλον. Η Ευρώπη δεν έχει κάνει πολλά για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και την ιστερία. Ε, κανείς δεν αρνείται ότι είναι μια κρίση αυτή, όμως είναι μπροστά σε μια κρίση η Ευρώπη πρέπει να κατήσει την ψυχραιμία τη. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αγνοούμε τις ε, παραπλανητικές εξαρτίες ε, πληροφόρηση. Θα πρέπει εμείς να δίνουμε συγκεκριμένες ε, τακτικές πραγματικές πληροφορίες και αξιόπιστε πληροφορίε στους πολίτες μας η εμπιστοσύνη τους είναι το πιο πολύτιμο αγαθό και η παραπληροφόρηση είναι ίσως κάποιες φορές ακόμα πιο μεταδοτική από ότι ο ίδιο ο κορονοιό. Σας ευχαριστώ ο κύριος Πουτικόφερ τώρα, εξ ονόματος των Πρασίνων. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τον κινέζικο λαό και ειδικά τους ανθρώπους του Γουχάν. φρυνούμε για τα θύματα και συλληπόμαστε τους οικείους των νεκρών. Εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος ε, την δουλειά που κάνουν ε, οι Κινέζοι οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή υπό πολύ ψηλού κινδύνους και θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερος το θάρρος και την αυτοθυσία του ιατρού Λιγουνιάν και των υπολείπων. Καλωσορίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, έδειξαν με κάποιες πρώτες αντιδράσεις στήριξης της Κίνας. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε συνεργασία και βοήθεια. Η κρίση αυτή δεν έχει περάσει. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια εντός της Ένωσης και ειδικά μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό στηρίζω πλήρως τα όσα είπαν οι συνάδελφοι πριν. Γενικά έχει σημασία η διεθνή συνεργασία. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως το ότι η Ταϊβάν πρέπει να περιληφθεί στις ε, προσπάθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και τέλος, υπάρχει μια βαθύτατη ανησυχία και ευχαριστώ την κυρία Επιτροπό που το ανέφερε για τις ε, αναφορές περί ξενοφοβικών περιστατικών σε κάποιες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατά Κινέζων ή Ασιατών. Είναι απολύτως απαράδεκτο. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη και όχι ξενοφοβία και ρατσισμό. Και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσει ε, και την διασπορά τους. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κόπτσινσκα από το mm, ECR. Ευχαριστώ. Λαμβάνοντας υπόψη το επίγον του προβλήματος, έχω δύο ερωτήσει να θέσω στην Κομισιόν. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για το, την αυριανή έκτακτη συνεδρία... των Υπουργών Υγείας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης ε, Ασθενειών συντονίζουν τις ενεργεία τους. Και θα μπορούσε επίσης να μας πει η Κομισιόν πότε θα εκδώσει το, την πέμπτη αξιολόγηση κινδύνου Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς συντονίζετε τη δράση σας με τρίτες χώρες. Ιδιαιτέρως έχετε σκεφτεί να ληφθούν εκτακτά μέτρα στην περίπτωση που ο ιός διαδοθεί πολύ στην Αφρική, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα τα συστήματα υγείας των χωρών της Αφρικής ο Γενικό Διευθύντη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία είπε ότι μπορεί να μην διαθέτουμε εμβόλιο για τους επόμενου 18 μήνες. Έχετε παρόμοια αξιολόγηση εσεί. εκτίμηση μάλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σουρμπάν Κρέσπο, μέρο τη ΓΚΟΕ. Ο κορονοϊός ε, είναι λιγότερο θανατηφόρος από μια συνήθη γρήπη, αλλά η, ο πανικός είναι πολύ πιο ισχυρός. Ε, τα στερεότυπα μάλιστα δημιουργούν και επιτείνουν διακρίσεις εναντίον των Ασιατών. Ο ιός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ρατσισμό, αλλά με βελτίωση ε, της πρόσβασης σε καθολικά και δωρεάν συστήματα υγείας καθολική πρόσβαση συστήματα υγεία είναι θεμελιώδης δικαίωμα και τα μέτρα λιτότητας θα πρέπει να αντιστραφούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στα συστήματα υγεία και η ποιότητα των συστημάτων υγεία. Η διαχείριση τέτοιων κρίσεων θα πρέπει επίσης να γίνεται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλο, απαιτούμε να εστιάσουμε στην μηδενική ανοχή ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον ατόμων ασιατικής προέλευσης. Γιατί αυτό είναι ο κίνδυνος και όχι τόσο ο ιός. Ο κ. Στέφανης τώρα, εκ μέρους του ΕΛΚ. Όπως... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ήδη γνωρίζουμε, Ήδη υπάρχουν χίλια θύματα του κορονοϊρού και 440.000 ε, άνθρωποι που έχουν μολυνθεί με τον ιό. Ε, επίσης, ε, η Κίνα δεν συμμετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις ε, του ΠΟΗ. Η Ταϊβάν είναι ο πιο το πιο σημαντικό κόμβος ε, ε απενδυτικός στην Νοτιοανατολική Ασία και είναι καιρός να συνεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε. Ε, γι' αυτό σας ζητώ, συνάδελφοι, να στηρίξετε την κοινή μας έκκληση για όλους όσους εργάζονται ε, στους ε, διεθνείς οργανισμούς. Η Ταϊβάν θα πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μπορούμε να, να νικήσουμε αυτήν την ε, τρομακτική αρρώστια μόνο συνεργαζόμενοι όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να αποτρέψει την διάδοση του ιού αλλά και τη διάδοση της προπαγάνδας που σχετίζεται με τον ιό στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά μέσα. Οι Κομισιόν και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εγκρίνουν τα σχετικά μέτρα. Πολλά πράγματα έχουν γίνει, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Ξέρουμε ότι υπήρχαν λίγα μεμονωμένα κρούσματα στην Ευρώπη. Και πρέπει να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Να ενημερώσουμε. Να δοθεί έμφαση στην πρόληψη, η οποία είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Επίσης να επισημάνω ότι υπάρχει έλλειψη μασκών εξαφανίζονται από την αγορά. Πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι η αρρώστια αυτή μεταδίδεται και από τα μάτια, τις μύτες και το στόμα. Απευθύνω λοιπόν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να διαδοθούν οι σχετικές πληροφορίες προς πολίτες. Σας ευχαριστώ. Τριλέ Λενουάρ για το Ρινιό. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή. Ο κορονοϊός μας οδηγεί σε παγκόσμια κρίση γιατί δεν εμποδίζεται από τα σύνορα. Η Κομισιόν πολύ σωστά παίζει το ρόλο του συντονιστή μεταξύ των κρατών μελών, εκδίδει συστάσεις για το ιατρικό προσωπικό, βοηθάει στην, στον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών από την Κίνα, χρηματοδοτεί έρευνα με 10 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αναζητηθούν καινούρια φάρμακα και εμβόλια. Ακούσαμε τα τελευταία, τις τελευταίες μέρες ε, πολύ κριτικές, επικριτικές ε, ε, γνώμες για την κινέζικη κυβέρνηση. Δεν, το πρόβλημα δεν είναι να δείξουμε το δάχτυλο κάποιον, ούτε να χρησιμοποιήσουμε την περίπτωση αυτή για ιδεολογική διαμάχη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε το ιατρικό προσωπικό και την κυβέρνηση Κίνας να αγκαλιάσουμε να, τις ε, χώρες της Αφρικής επίσης που έχουν πολύ ευαίσθητα συστήματα υγείας και δεν θα επιτρέψουν ε, να περιοριστεί η επιδημία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο ε, στην επόμενη ομιλήτρια, ε, να ανακοινώσω ότι έχουμε πέντε υποψήφιους για το Catch the Eye. Θα λάβουν και οι πέντε το λόγο, αλλά κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών στο Catch the Eye. Ε, ο λόγος τώρα στην κυρία Ντεσούτερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καμία χώρα μόνη της ε, δεν μπορεί να σταματήσει την επιδημία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη, την κινέζικη κυβέρνηση και άλλους εταίρους. Και την Ταϊβάν. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για να σταματήσει η επιδημία. Αλλά δεν πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να πέσουν και αυτά θύματα του ιού. Πολλέ οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν πει πω η κινέζικη κυβέρνηση αποκρύπτει πληροφορίε. Και δεν επιτρέπει πρόσβαση σε τρόφιμα και φάρμακα. Αλλού υπάρχει αύξηση της αντικινεζικής ξενοφοβίας. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Σε περιπτώσεις ε, δημοσίας ε, υγείας οι περιορισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι αναλογικοί, να βασίζονται στην αναγκαιότητα και στα μέτρα που χρειάζονται να προστατεύσουμε την υγεία μας. Αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το ΕΛΚΟ κύριος Λίζε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους συγκινείς των νεκρών και εγώ στηρίζω τα όσα είπα η Επίτροπος ότι πρέπει να συνεργαστούμε στην Ευρώπη. Αλλά αν βλέπουμε στον τίτλο της συζήτησης τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να πούμε πως ε, εδώ πέρα ο περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης οδήγησε σε επιδείνωση της κρίσης. Και ένα κομμάτι της παγκόσμιας κοινότητας η Ταϊβάν έχει αποκλειστεί για ιδεολογικούς λόγους από το συντονισμό και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι ένα σημαντικό μήνυμα απόψε. Η ιδεολογία δεν μπορεί να είναι πάνω από την υγεία. Αυτό και στην Κίνα νομίζω πρέπει να γίνει σαφές. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φριτσόν για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτροπέ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Ο κορονοϊός έχει ανησυχήσει όλο τον κόσμο. Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πολύ τις τελευταίες μέρες. Και είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να δίνουν, να παρέχουν συνεχώς ε, ορθές πληροφορίες ε, στους πολίτες. Προφανώς είναι κρίσιμη σημασία και η έρευνα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η θέση σε καραντίνα των υπόπτων ε, θα λαμβάνει χώρα αλλά δεν θα παραβιάζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα των επιθέσεων εναντίον ατόμων που μοιάζουν με Ασιάτες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη διάδοση του ιού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ντάλη που ξεκαθάρισε τις ευθύνε της Κομισιόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Βίσλερ Λίμα από το ΕΛΚ. Ε, ο Λίου Αλιάνγκ ήταν ο γιατρός ο οποίος είχε προειδοποιήσει για τον ιό και αν τον είχαμε ακούσει θα είχαμε περιορίσει τον ιό πολύ νωρίτερα. Όμως οι αρχές στην Κίνα ε, τον κατηγόρησαν ότι ε, απειλούσε την ε, δημόσια τάξη. Αν είχε εισακουστεί τότε ο γιατρός αυτός, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε. Η διαφάνεια σε θέματα υγείας θα πρέπει να επικρατεί πάντοτε, όπως και η κοινή λογική. Θα είχε επιτρέψει αυτό, θα έπρεπε να επιτραπεί η Ταϊβάν να συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο γιατρός Λι Βαν δυστυχώς πέθανε. Θα έπρεπε το όνομά του να αποτελέσει συνώνυμο της έκκλησης για την ελευθερία του λόγου. Ε, αυτή τη ε, στιγμή πολλοί άνθρωποι ε, φυλακίστηκαν επειδή ενημέρωσαν την κοινή γνώμη μέσω των μέσων κοινωνική δικτύασης για κρούσματα ε, και γίνεται μια προσπάθεια συγκάλυψης. Ε, θέλω εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται χωρίς ξεκούραση για την καταπολέμηση του ιού. Έχετε μια μπλε κάρτα, λέει η Πρόεδρος. Τη δέχεστε? Oui? Yes, sure. Okay. Μάλιστα. 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε διαβάσει ε, το βιβλίο La Peste του Αλμπέρ Καμιν. Ναι, και στο τέλος αυτού του βιβλίου η τελευταία φράση λέει ότι ο ιός ε, δεν πεθαίνει ποτέ και θα πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί. Ο Καμίου λέει ότι η ελευθερία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντοτε να προστατεύουμε. Ε, στο βιβλίο αυτό έκανε λόγο για την μαύρη πανόλη. Ε, και η, ε, οι θεμελιώδεις ελευθερίες τις οποίες στην πραγματικότητα αναφέρεται είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατεύουμε πάντοτε. Χαίρομαι που μιλήσατε για αυτό το βιβλίο La propia... Queremos cerrar. η... η Κίνα αντιμετώπισε τον ιό με πολλές αδυναμίες ε, και χωρίς διαφάνεια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στην Αφρική. Ε, όλα τα συστήματα υγείας υφίστανται πιέσεις εξαιτίας του ιού και θα, υποστούν και στο μέλλον. Ε, για παράδειγμα, τη μεγάλη ε, έκθεση για τα κινητά τηλέφωνα της Βαρκελόνης ακυρώθηκε σήμερα το απόγευμα εξαιτία μειωμένη συμμετοχής. Τι ζητάμε. Ζητάμε μια ενιαία συντονισμένη αντιμετώπιση με όλα τα κράτη-μέλη. Μια στρατηγική, κοινή στρατηγική επικοινωνίες που θα καθησυχάζει και θα διασφαλίζει τη ζωή όλων των Ευρωπαίων. Μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε ε, τα, τις, ψευδείς, τις ειδήσει και το στίγμα. Εγώ ως πολίτης πραγματικά θα ήθελα να διαθέτω στα κέντρα υγείας πληροφορίες για το πώς μπορούμε να προλάβουμε τον κορονοϊό. Εμείς λοιπόν πρέπει, πρέπει να πάρουμε μέτρα με μια συγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνία, συντονισμό, συντονισμένη, ε, να διαθέτουμε στοιχεία ε, μέσω ερωτηματολογίων που δίνουμε στους εισερχόμενους επιβάτες και με συντονισμό με τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε αύριο πετούμε από τους Υπουργούς Υγείας και από την Επίτροπο να δώσουν μια ενιαία και συντονισμένη απάντηση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σταγιάννη έχει τώρα το λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι σαφής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο είναι σαφή. Εμεί στηρίζουμε τη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τη ζητάμε από αύριο το πρωί να ε, προσπαθήσει να δώσει συντονισμένη απάντηση από πλευρά όλων των κρατών μελών τη Ένωση, ενωμένη με τα ίδια μέτρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια επίγουσα κατάσταση που δραματικά χτύπησε την Κίνα και δεν θέλουμε να χτυπήσει και την Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται ενότητα, χρειάζονται μέτρα. Εμείς προτείναμε το, ένα ερωτηματολόγιο που επιτρέπει να καταλάβουμε αυτοί που φτάνουν στην Ευρώπη αν έχουν περάσει στην Κίνα ε, σε περιφέρειες όπου ε, έχει ε, διαδοθεί η, ε, η αρρώστια. Να μην ε, δράσουμε με πανικό, να δράσουμε συντονισμένα. Η Κίνα τέλος δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και συνεχίζει να μην κάνει αυτά που πρέπει. Δηλαδή μας δίνει λοιπέ πληροφορίε, ξεκίνησε καθυστερημένα. Οι Κινέζοι είναι το πρώτο θύμα ενό συστήματο που έκανε όπω έκανε και η Σοβιετική Ένωση με την υπόθεση του Τσερνομπίλ. Κρύβει τι τραγωδίε και σημαίνει αυτό πρόκληση τεράστιων ζημιών στου ίδιου του πολίτε τη. Οι Κινέζοι είναι τα πρώτα θύματα του κομμουνιστικού καθεστώτο τη Κίνα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε την διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Τσοχαντάρου είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη στιγμή που μιλάμε, ο αριθμός ε, των θυμάτων έχει φτάσει έχει πολλαπλασιαστεί επί χίλια από την πρώτη φορά που εμφανίστηκε η, ε, ο ιός ε,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 όλοι πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή, άσχετα από τι πολιτικέ μα πεπιθήσει. Εγώ ήμουν υπέρ εξ αρχή ενό ολοκληρωμένου συστήματος δράση, ε, τον ενεργοποίηση του μηχανισμού έγκαιρη προειδοποίηση κτλ. Όλα αυτά τα μέτρα είναι καλά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε. Εάν χρειαστεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε πώ δεν έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές όσον αφορά τα συστήματα υγεία στα κράτη-μέλη μα και νομίζω πω θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια ε, ομοιόμορφη αντίδραση. Ελπίζω πως αύριο το πρωί, επίτροπε, ε, θα έχετε ε, ήδη ένα σύστημα ολοκληρωμένης αντίδρασης για τα θέματα υγείας και να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε. Και όπου εγώ ε, ε, έδρασα εθελοντικά για το έμπολα, γιατί είμαι επιγοντολόγος στη Ρουμανία, είμαι γιατρός, έτσι θα ε, ε, προτείνω ο ίδιος τον εαυτό μου εθελοντή και για την αντιμετώπιση αυτής της ε, κατάστασης. Ευχαριστώ παρακαλώ. Τελειώνει ο χρόνος μας. Κυρία Ντάλη, ένα λεπτό μόνο. Ακριβώς ένα λεπτό. Ευχαριστώ πράγματι. Στην Ελλανδία έχουμε πάνω από 2.000 ανθρώπου, θανάτους λόγω του κρύου και της ε, φτώχειας. Αυτός ο ιός έχει οδηγήσει σε πάνω από χίλιους θανάτους. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε μια αίσθηση της προοπτικής. Ο Επίτροπος είπε να το αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό οι επιστήμονες, να τονίσουμε την έρευνα, τις ε, κλινικές δοκιμές, το περιορισμό και τη συνεργασία. Εγώ θέλω να χαιρετήσω την προσπάθεια των Κινέζων που έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να περιορίσουν αυτή την επιδημία υπό δύσκολες συνθήκες και νομίζω πως όλα τα κρατη πρέπει αντίστοιχα να λειτουργήσουν και να διπλασιάσουν τι προσπάθειε του. Ο επίτροπο, είπε πω τα κατημέλια έχουν εισάγει διάφορα μέτρα στα σημεία εισόδου τη Ένωση. Θα πρέπει να πω ότι στη χώρα από την Ιρλανδία δεν έχουμε κάνει και πολλά, αλλά καλωσορίζω τι πατρίσει. σα πρέπει να βοηθηθεί η Κίνα, είναι σημαντικό αυτό και να ε, ε φροντίσουμε κατά των διακρίσεων γύρω από αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. επόμενο ομιλητή, κυρία Σόιντροβα από το ΕΛΚ. Yes. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Ε, συμφωνώ με πολλούς από τους προλαλήσαντες. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική, το ίδιο και η ευαισθητοποίηση. Οπότε δεν καταλαβαίνω πώς η, Κίνα η οποία ε, θέλει, ζητά συνεργασία, έχει αρνηθεί τη βοήθεια της ε, Ταϊβάν. Ε, το σύστημα υγείας της Ταϊβάν είναι ένα από τα πιο προοδευμένα, πιο επιτυχημένα στον κόσμο και θα έπρεπε μάλιστα η Ταϊβάν να εκπροσωπείται και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η υγεία υπερβαίνει την πολιτική, κατά την άποψή μου. Θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να εξασφαλίσετε ότι να πιέσετε την Κίνα να σταματήσει να αρνείται τη βοήθεια της Ταϊβάν. Εμείς είμαστε υπέρ της αλληλεγγύης, οι ε, πολίτες αυτή τη στιγμή στην ε, Τσεχία ε, στέλνουν χρήματα στην Κίνα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ ο κ. Ζαχραντήρ από το ECR. Χαίρομαι που ακούω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη και πρόθυμη να αντιμετωπίσει αυτή την επικίνδυνη πανδημία και χαίρομαι που θα συνεργαστείτε με την ε, Κίνα. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι στρατηγική συμμαχία από το 2003 και έχουμε δει μάλιστα και αποτελέσματα, ε, ε, θετικά αποτελέσματα από τότε στην οικονομική ανάπτυξη. Τώρα όμως έχει χτυπηθεί από αυτή την ασθένεια και μπορεί και αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναζωογονήσουμε αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση. Όπως είπε ο κ. Μπουτικόφερ προηγουμένως, πρέπει να συμπεριλάβουμε καλύτερα την Κίνα στο πλαίσιο δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και προφανώς να αντιμετωπίσουμε και κάποιες συμπεριφορές εναντίον των Ασιατών και εναντίον των Κινέζων υπηκών που διαδίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριος έχει το λόγο. One minute. Would I dare take any... Ε, εντάξει, δεν θα μιλήσω παραπάνω από ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το 2009 είχαμε την γρήπη των χείρων στις ΗΠΑ. Ξαπλώθηκε σε 100 χώρες. Πάνω από 10.000 άτομα πέθαναν. Φέτος μόνο στις ΗΠΑ 19 εκατομμύρια άνθρωποι αρρώσαν από γρήπη, 10.000 πέθαναν. Είναι διασκεδαστικό το πώς έχει χρησιμοποιηθεί το θέμα αυτό για να υπονομευτεί το κινέζικο κράτος. Και είναι και τρομακτικό. Αν ε, έχουν πρόβλημα με τον κορονοϊό οι Κινέζοι δεν χρειάζονται τη βοήθεια και τη συνεργασία μας. Δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε και να τους χτυπάμε. Έχθεσαν ένα νοσοκομείο σε δέκα μέρες. Εμείς ούτε τη χαρτούρα δεν θα κάναμε σε έξι μήνες. Το κράτος τους ήταν έτοιμότερο από πολλά άλλα για να αντιμετωπίσει την κρίση και πρέπει να τους ε, χειροκροτήσουμε. Ο ήταν, θετικό, ο ΠΟΕ ήταν θετικός για την αντίδρασή τους, αλλά Τώρα να μιλάνε οι Ευρωπαίοι και να λένε για ανθρώπινα δικαιώματα και τέτοια για να υπονομεύσουν τους Κινέζους ε, είναι πραγματικά απίστευτο. Έχουμε πολλά να διδαχτούμε από τους Κινέζους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ανταλή να απαντήσει. Πατήστε το μικρόφωνο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές για την ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Σημείωσα όλα σας τα σχόλια. Όσον αφορά την Ταϊβάν, για το σε ποιον ακριβώς προωθούμε πρακτικές λύσεις χωρίς την συμμετοχή της Ταϊβάν στο διεθνές πλαίσιο. Ε, αυτό γίνεται, είναι συμβατό με την πολιτική της μίας Κίνας. Όσον αφορά τις κινέζικες υπηρεσίες, είμαστε σε καθημερινή επαφή και δεν έχουμε κάποιον λόγο να αμφιβάλλουμε για τις πληροφορίες που μας δίνουν. Επίσης, ε, να σας πω πως είμαστε σε επαφή με τις Αφρικανικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια συμφωνία συνεργασίας με το Κινέζικο Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών. Φροντίζουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, οπότε δεν χρειάζεται πανικός, αλλά επαγρύπνηση. Οπότε, εκτιμώ το ότι έχουμε ένα κοινό στόχο εδώ, να διασφαλίσουμε μια ενιαία αντίδραση στην επιδημία αυτή. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε. Όμως η επιτυχία εξαρτάται και από την συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή όλων των μέρων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως σήμερα είδαμε εδώ πέρα την πολιτική βούληση που υπάρχει. Θα υπάρξει λοιπόν αύριο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας και θα έχουμε άλλη μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσουμε τον συντονισμό μας. Απαιτείται επίσης να ευθυγραμμίσουμε τα μέτρα ετοιμότητας και αντίδρασης και στα εξωτερικά σύνορα. Έτσι θα στηριχθούν οι προσπάθειες της ε, Κίνας για να περιοριστεί ο ιός ε, και να μην διαδοθεί άλλο εντός της Ένωσης, αλλά και για να βοηθήσουμε τρίτες χώρες. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, να στηρίξουμε την Κίνα και την διεθνή αντίδραση. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του συνεγγύς θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και οπωσδήποτε θα ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνεδρίαση θα επαναληφθεί αύριο το πρωί σε 9. Η ημερήσια διάταξη υπάρχει στη σελίδα του Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ.